Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Συνεχίζει τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να ανακοινώσω το αποτέλεσμα για την υποψήφια 16 υπέρ 2 κατά 2 εποχές με το διορισμό της ε, κυρίας Γκαλπέλ στο ελεκτικό συνέδριο. Προχωρούμε. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω την κυρία Ιβάνοβα για την ειδική έκθεση 5 του 2017 από το ελεγκτικό συνέδριο. Please take your seat. We need to go ahead. And if you want to discuss, leave. Παρακαλώ, πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση και αν θέλετε να ε, συζητήσετε εκτός έθους. Έλεγα λοιπόν η ειδική έκθεση 5-2017 για την εγγύηση για την νεολαία και τις ευρωπαϊκές πολιτικές κατά πόσο βοήθησαν την απασχόληση. Κυρία Ιβάνοβα, καλώς ορίσατε. Σας δίνουμε αμέσως το λόγο. Και μάλλον θα σας ε, ενισχύσει, θέλουμε ενισχύσεις και άλλη γυναίκα στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχετε αμέσως το λόγο. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντοτε με χαρά βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ και για την ευελιξία σχετικά με την παρουσίαση αυτής της ε, έκθεσης μόνο λίγες μέρες μετά τη δημοσίευσή της στις 4 Απριλίου. Να συγχαρώ τον κύριο Βόν, τον εισηγητή, για ένα πληρέστατο έγγραφο εργασίας ε, το οποίο προετοιμάσει δεδομένης και της περιπλοκότητας και της ε, πληθώρας δεδομένων. Η ανεργία των νέων είναι μία από τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 2013, αλλά άνω των 4 εκατομμυρίων, 4,2 είναι ακόμα άνεργοι ήταν στα μέσα του 2016 με μέσο ποσοστό 18,8%. Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι αυτών των μεγάλων περιόδων ανεργίας είναι πολύ αρνητικός και για την μελλοντική απασχολησιμότητα και για τον κοινωνικό αποκλεισμό και γενικά για τη χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Το σημείο κίνησής μας ε, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε αυτή την τρίτη κατά σειρά έκθεση που αφιερώνεται στο θέμα της ενεργείας μεταξύ των νέων, κοιτάξαμε δείκτες μεταξύ των ε, δεδομένων ΕΜΚΟ, την εξέλιξη πέραν της εκπαίδευσης και της κατάρτασης, της ε, καταχώρησής τους, των, της προσφοράς που υπάρχει και της βιωσιμότητας των προσφορών αυτών, για απασχόληση δηλαδή. Ελέγξαμε επίσης κατά πόσο τα κράτη-μέλη καλύπτουν τους ε, επιπρόσθετους παράγοντες που διαμορφώνουν την ενεργεία των νέων και τους στόχους ε, του εγγυητικού μέσου για τους νέους. Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβακία εξετάσαμε στα πλαίσια της έκθεσης, της μελέτης, επί τη βάση μιας σειράς κριτηρίων, όπως η ενεργεία των νέων, οι ανάγκες επί του συνόλου του πληθυσμού και το μερίδιό τους στις συνολικές κατανομές των κονδυλίων. Συνολικά το συμπέρασμά μας είναι ότι τα 7 κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε αυτά πράγματι είχαν σημειώσει κάποια πρόοδο με την υλοποίηση του εγγυητικού μέσου για τους νέους και είχαν επιτευχθεί κάποια αποτελέσματα, αλλά κανένα από τα κράτη-μέλη αυτά δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει προσφορά εντός τεσσάρων μηνών. Και είχαμε πολύ περιορισμένη επιτυχία σε σχέση με τους στόχους που είχε διατυπώσει το μέσο. Ως προς τα δεδομένα για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και τις διάφορες φάσεις που βρίσκεται το κάθε κράτος ε, για την ταυτοποίηση και καταχώρηση της οποιασδήποτε προσφοράς απασχόλησης, θα εστιαστώ μόνο σε κάποια πορίσματα, σε κάποια από τα πορίσματά μας. Εδώ είχαμε αποτελέσματα στοχευμένα εξ αρχής, αλλά η αύξηση του πληθυσμού των νέων είχε σχέση, των ανέργων νέων δηλαδή, είχε σχέση και με την αύξηση του συνολικού πληθυσμού των νέων. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας δεν αυξήθηκε με την εισαγωγή του μέσου του εγγυητικού, αλλά δεν είχαμε επαρκή αριθμό προσφορών και το 70% εκείνων που εκμεταλλεύτηκαν τέτοιες προσφορές το έκανε εντός τεσσάρων μηνών, αλλά η αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασία των ανθρώπων αυτών παραμένει προβληματική. Για τα 7 κράτη-μέλη βρήκαμε ότι μόνο το 48% των νέων που ολοκλήρωναν το εγγυητικό μέσο το 2015 ήταν ακόμα απασχολούμενοι σε πρόγραμματα κατάρτιση εκπαίδευση μετά από 6 μήνες. Αναλύσαμε επίσης τους παράγοντες που επιδρούν ε, επί των αποτελεσμάτων αυτών και βρήκαμε τους κυριότερους λόγους για τα περιορισμένα αποτελέσματα. Έλλειψη δηλαδή σαφών στρατηγικών με σαφή σημεία ε, συγκριτικής ανάλυσης, αξιολόγησης. Ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη στόχευσαν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και απέκλεισαν ευθύς εξ αρχής με τα κριτήρια που έθεσαν τουλάχιστον το 30% του συνολικού πληθυσμού. Επίσης δεν υπήρχε επαρκής εκτίμηση του κόστους και της υφισταμένης ε, χρηματοδότησης. Η προσέγγιση των κρατών μελών επίσης επιδρά επί της αποτελεσματικής ε, ένταξης των αναγκών. Σε κάποιο βαθμό η ποιότητα των δεδομένων ήταν εμπόδιο. Και η τρίτη πτυχή που είναι πολύ σημαντική έχει σχέση με την συνεισφορά της πρωτοβουλίας ή στα πλαίσια του μέσου του εγγυητικού Εκεί έχουμε κάποια προβλήματα λοιπόν σχεδιασμού και προγραμματισμού και ένας κίνδυνος τα κονδύλια EASF e να αντικαταστήσουν τα εθνικά κονδύλια στις περιοχές αυτές. Και εδώ οι κατευθύνσεις κομισιών για την συλλογή δεδομένων επιδρούν επί της επιμέτρησης και η πρόχρηματοδότηση για τα κονδύλια EASF e δεν έγινε με απόλυτα αποτελεσματικό τρόπο και τα μέτρα που υποστηρίχθηκαν από η ΑΕΕ η ESF ε, υποπαρέδωσαν για να το πούμε έτσι. Αυτοί που περισσότερο εκμεταλλεύτηκαν ε, τα συγχρηματοδοτούμενα μέσα ήταν εκείνοι με τους οποίους, όχι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά εκείνοι με τους οποίους μπορούμε πιο εύκολα να έρθουμε σε επαφή. Επομένως οι προσδοκίε του εγγυητικού μέσου δεν έχουν καλυφθεί. Έχουμε κάποιες βελτιώσεις και κάποια πρόοδο, τη δημιουργία δηλαδή συστημάτων παρακολούθησης, τον ορισμό μια καλής προσφοράς, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ή του ελλείμματος δεξιοτήτων και εδώ έχουμε και μια σειρά από συστάσεις 7 στον αριθμό που απευθύνουν τα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν η πιο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση των προσδοκιών, θέτοντας ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους. Επίσης, η συνολική εικόνα του κόστους του εγγυητικού μέσου σε σχέση με την υφιστάμενη χρηματοδότηση. Ε, στην ουσία, αυτή είναι η αιστεία της εκθέσεως Προφανώς γνωρίζετε όλοι ότι στις 10 Μαΐου έχουμε μια υψηλού επίπεδου συνεδρία, συνέδριο. Η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Και είμαι έτοιμη εδώ να ακούσω τις, τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you for your presentation. You have... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Θα παρατηρήσατε ότι η πρόεδρος κυρία Γκρέσλε αποχώρησε για λίγα λεπτά μόνο, οπότε θα προεδρεύσω και θα παρουσιάσω και το έγγραφο εργασία μου. Απλά καφέ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα φτιάξω. <laughs> να ξεκινήσω λοιπόν ε, ευχαριστώντα σα για την έκθεση και για τη διοργάνωση της ε, διάσκεψης τη 10ης ε, Μάιου. Θα συμμετέχουμε και νομίζω ότι μόνο και μόνο το ότι οργανώνεται αυτή τη διάσκεψη δείχνει τη δέσμευση που έχετε αναλάβει και το πόσο σημαντικό θεωρείτε το θέμα αυτό για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Θα ήθελα λοιπόν να, κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και περνάω μετά στις συστάσεις μου. Οι γενικές παρατηρήσεις ε, ήταν και δική σας αφετηρία και η δική μου αφετηρία είναι ότι πάντοτε στηρίζω το σχήμα για τις εγγύσεις, για την νεολαία και τη χρηματοδότηση γιατί θεωρώ ότι η ανεργία των νέων είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής μας. Αν δείτε τα νούμερα σε ορισμένα κράτη-μέλη, πραγματικά αποτελεί ντροπή, όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο η ανεργία των νέων είναι 18% ε, και σε πολλά κράτη βέβαια πολύ παραπάνω από αυτό. Ε, πρέπει να πω ότι ήταν μια πολιτική απόφαση η δημιουργία της εγγύης για την νεολαία και ήταν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και πολλά κράτη δεν είχαν ε, την ε, δομή έτοιμη ε, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα σχήματα αυτά των εγγύσεων για την ολια Σιγά σιγά ξεκινάει και έχει πάρει και κάποια ρυθμό η προσπάθεια αυτή παρότι ξεκίνησε αργά. Το θέμα είναι να γνωρίσουμε τα δεδομένα ε, που είναι από το 2014-2015, οπότε και πρωτοξεκίνησε η πρωτοβουλία ε, της εγγύησης για την νεολαία και του EA. Και βέβαια νομίζω ότι σωστό είναι να πούμε ότι το σχήμα αυτό, το πρόγραμμα εγγύσεων για την νεολαία, έχει βοηθήσει χιλιάδες νέους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει αυτό να το ξεχνούμε. Και πραγματικά έδωσε ευκαιρίες σε πολλούς νέους ε, η αφετηρία μου λοιπόν είναι ότι όταν θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίε ε, για τους νέους, αυτές οι ευκαιρίε θα πρέπει να είναι και ποιοτικέ. Δεν μπορούμε απλά να δίνουμε κάτι ε, στους νέους, απλά για να τους βγάλουμε από τα μητροανέργων. Οποιαδήποτε ευκαιρία, θέση εργασία ε, ή θέση ασκούμενου πρέπει να είναι ποιοτική θέση για να μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτήν οι νέοι και να για το μέλλον του. Είδατε, είδαμε μάλλον ε, την έκθεση και τις συστάσεις του ελληνικού συνεδρίου, ε, ακούσαμε και είδαμε και τι λέει η Κομισιόν. Δεν είναι 100% ικανοποιημένη η Κομισιόν. Τα δέχονται σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τη έκθεση που αμφισβητούν. Φαντάζομαι θα μα τα πει και εκπρόσωπος, ή η εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή αργότερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι δικέ μου συστάσει, ε, φαντάζομαι ότι τι έχει διαβάσει και δεν θέλω να ευσέλθω σε λεπτομέρειε μειώνεται η ανεργία των νέων παρότι παραμένει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είπα παραμένει το ποσοστό υψηλό 18% κατά μέσο όρο. Πρέπει όμως να παραμείνει γι' αυτό το λόγο προτεραιότητα η καταπολέμηση ανεργίας των νέων και να βρούμε τρόπους ε, είτε με τον οργανισμό για την απασχόληση των νέων, είτε με, τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν στα προγράμματα εγγύσεων για την νεολαία και να περιμένουν μόνο από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Επίση, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Στην έκθεσή σα και στην προφορική σα σήμερα παρουσίαση αναφέρατε το ότι κανένα από τα κράτη-μέλη που επισκεφθήκατε δεν μπορούσε να πάρει μια προσφορά εντό τεσσάρων μηνών από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία Άρα μεγάλο μέρος ευθύνης ε, είναι στα κράτη-μέλη και πρέπει να υπάρξουν σωματικές βελτιώσει στο μέλλον. Ε, το είπα και στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό η προσφορά να είναι ποιοτική. Στην έκθεσή σας μου αρέσει η αναφορά το να αντιμετωπίσουμε την αναντιστοιχεία δεξιοτήτων. Πραγματικά χρειαζόμαστε πληροφορίες ε, για την αγορά εργασίας, ώστε η κατάρτιση που προσφέρουμε στους νέους να είναι πράγματι χρήσιμη για αυτούς, να μπορούν να βρουν δουλειά. Και στη δική μου χώρα και αλλού βλέπουμε ότι εκπαιδεύουμε τους νέους για να τους βγάλουμε από τα μητρώα ανέργων, απλά και μόνο γι' αυτό όμως, χωρίς να τους δίνουμε εφόδια για να μπορούν να βρουν μια δουλειά στην αγορά εργασίας. Αυτές είναι βασικά οι δικές μου συστάσεις. Και αν μου επιτρέπετε, έχω και κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φαντάζομαι σε λίγο θα λάβουν το λόγο οι πρόσωποι. Πρώτη ερώτηση προς την Κομισιό. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα προγράμματα αγγίση για την νεολαία ε, παρακολύθηκε από την έλλειψη πόρων. Έχουμε αυτό τον προπολογισμό 6,4 δις. Ε, επαρκεί ή χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση για να υποφεληθούν από αυτό το ε, πρόγραμμα εγγύησεων περισσότεροι νέοι. Επίσης, μπορεί να μας πει η Κομισιόν τι βελτιώσεις θεωρούν ότι έχουν ήδη γίνει μετά την έκθεση του εκλεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος βάλει πρώτο στον κατάλογο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και την πολλή δουλειά που έκανε για το εγγυητικό μέσο για την νεολαία είχαμε την ευκαιρία από κοινού να διαπιστώσουμε την κατάσταση στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μαζί με την συνάδελφο Νταλαμπαγιόβα. Εμείς σημειώσαμε λοιπόν τα της του μέσου στην Ιταλία και διαβάζοντας και τις συστάσεις νομίζω του ελεγκτικού συνεδρίου θα έλεγα ότι συμφωνώ απολύτως και με τις τεχνικές και με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαδικασίες καταχώρησης των ενδιαφερομένων. προκειμένου να ενσωματωθούν δηλαδή στο μέσον. Θεωρώ ότι ε, το πρόγραμμα ε, του εγγυητικού αυτού μέσου δεν είναι μια απόλυτη αποτυχία. Κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η πολιτική τάξη βεβαίως που τα διαχειρίζεται, δεν ε, ήταν σε θέση να δημιουργήσουν μια δομή ώστε να απορροφήσει αποτελεσματικά και να διοχετεύσει αυτά τα κονδύλια που διατέθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν ένα πιο αυστηρό, πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα που να καταγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις ανάγκες των νέων και όλες τις λεπτομέρειες των όποιων καταβολών και της όποιας βοήθειας. Χρειάζεται επίσης να κάνουμε περισσότερη δουλειά ενημέρωσης προς τους πολίτες σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό. Ε, είδαμε επίσης ε, και κάποιες περιπτώσεις ε, προγραμμάτων λογισμικού προβλημάτων μάλιστα λογισμικού που καθυστερούσαν καταβολές προς τους δικαιούχους ε, νέους αρκετό χρονικό διάστημα ε, σε σχέση με ε, συμμετοχή σε προγράμματα στάζου, σε προγράμματα άσκησης. Αυτό έχει σχέση βεβαίως με θέματα οικονομικής διακυβέρνησης. Διότι το μέσο το εγγυητικό μέσο για τους νέους δεν μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ενημέρωσης και να βοηθήσει τα κρατημέλη να αναπτύξουν αντίστοιχες διαδικασίες ώστε οι νέοι άνεργοι να καταχωρίζονται στο πρόγραμμα και να βοηθούνται προς την ε, ε, έρευνά τους στην αγορά απασχόλησης. Χωρίς όμως μια ε, διαρθρωμένη στάσια της πολιτικής ηγεσία της κυβέρνησης σε κάθε χώρα ε, χωρίς να συνοδεύονται αυτά τα προγράμματα από μια ε, απλώς οικονομική λογική, ορθό λόγο. Δεν μιλάω για ιδιαίτερο θάρρος. Ε, χρειάζεται στις δημόσιες δαπάνες να κατευθύνουμε κάποια κονδύλια σε πολύ ευαίσθητου τομεί τη οικονομίας για την ε, ανάπτυξη. Ώστε όλα αυτά να είναι βιώσιμα, διότι διαφορετικά θα επανέλθουμε σε ένα σύστημα λογισμικό που να λειτουργεί θαυμάσια όπως το εγγυητικό μέσο, αλλά χωρίς αυτό να προσφέρει πραγματική βοήθεια στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό την μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή. Επομένως, πέραν των διατάξεων, των συνθήκων και τα λοιπά, των νομικών δεσμεύσεων, η δική μου σύσταση ε, είναι πολιτικής φύσεως. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι τεχνικές συστάσεις ε, είναι καλοδεχούμενες ε, και πολύ ενδιαφέρουσες και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις κυβερνήσεις που υλοποιούν τα προγράμματα αυτά. Ώστε το σύστημα να είναι πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό, να λειτουργεί, να επιτυγχάνει αποτελέσματα. Έτσι ώστε, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για ε, ασκήσεις νέων να μπορέσουν ενδεχομένως να κρατήσουν κάποιους από αυτούς τους νέους και να μην επανέλθουν αυτοί στην ανεργία που γνώριζαν προηγουμένω. προτού ενταχθούν δηλαδή στο πρόγραμμα ή στην οποιαδήποτε άσκηση. Μαθητεία. Να δημιουργούμε την ευκαιρία δηλαδή τελικώ της ένταξη στην ε, αγορά εργασία. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω κατά πόσον ε, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αυξηθεί το κονδύλι αυτό. Είναι, θα ήταν σωστό, εφόσον τα κράτη-μέλη σέβονταν τις συστάσεις και τις κατευθύνσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για να προσαρμόσουν τις διοικητικές του διαδικασίες. Γιατί βεβαίω είναι σωστή η αύξηση του κονδυλίου, αλλά υπό τι προποθέσει αυτέ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Λαβάγιο, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Ιβάνοβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλη την προσοχή που δίνετε στο θέμα αυτό, για την ενεργεία των νέων. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και χαρήκαμε που ήμασταν μαζί. Είχατε έρθει μαζί μας στην αποστολή στην Ιταλία και είδαμε η σώμαση, ε, ακριβώς τι συμβαίνει επί τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι που μας προκαλεί όλο και περισσότερα δεινά. Στην τσεχική δημοκρατία το ζούμε και υποφέρω εγώ πολύ, γιατί ε, βέβαια στην τσεχική δημοκρατία έχουμε ε, πολύ μεγάλο ποσοστό απασχόληση, καλύτερα και από τη Γερμανία. Αλλά σε άλλες χώρες ε, δυσκολεύτηκα, θα θυμάται ο Μπάρκο Βάλι πριν από ένα μήνα, όπου ένας νέος 22-23 ετών στην Ιταλία αυτοκτόνησε και είχε γράψει μια ανοιχτή επιστολή την οποία οι γονείς του δημοσίευσαν και κατηγορούσε ευθέως το σύστημα, την πολιτική, τους πολιτικούς και όλους εμάς ε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο, οφείλω να ομολογήσω, και οι χώρες αυτές που έχουν τόσο υψηλή ανεργία των νέων θα πρέπει να σκέφτονται το μέλλον τους και εμείς να αναρωτηθούμε, προβληματιστούμε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα, αν είναι χρήσιμα και αν μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των νέων μας για ε, το μέλλον. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι αρνητικές επιπτώσεις ε, και η μελλοντική απασχολησιμότητα και η ανάπτυξη οικονομική κτλ. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος για το ρόλο των νέων στην κοινωνία και στην Ευρώπη γενικότερα. Πάρα πολύ σοβαρό το θεωρώ αυτό το θέμα. Για την έκθεση σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετική η εργασία και ε, τα συμπεράσματά σας βασίζεστε στις πληροφορίες που συλλέξατε και για τις συστάσεις. Συμφωνώ απολύτως με όλες τις τεχνικές σας ε, συστάσεις. Θα πρόσθετα και κάποιες πολιτικές φυσικά εγώ και δεν θα πρέπει μόνο να βρούμε τα σφάλματα που πρέπει να διορθώσουμε, αλλά και να μάθουμε για το μέλλον, έτσι ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα. Δύο φορέ ίσως και περισσότερες, γιατί καμιά φορά σημαίνει και αυτό. Θα πρέπει να ε, δεσκόμαστε από τα σφάλματά μας. Και θα πρέπει να αναπτύξουμε και να ε, μοιραστούμε και καλές πρακτικές στην Ευρώπη. Το επαναλαμβάνω πάρα πολύ αυτό σε πολλές εκθέσεις. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητούμε για βέλτιστε πρακτικέ, τι χρησιμοποιούμε. Όχι. Τις αναφέρουμε σχεδόν σε κάθε έκθεση, αλλά δεν τις χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα. Γιατί δεν κοιτάμε τι κάνει καλύτερα ο γείτονα. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό και να το κάνουμε σε, μεταξύ των διαφόρων χωρών ακόμα και περιφερειών. Ευχαριστώ που το συνιστάτε αυτό. Επίσης θα πρέπει οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι και μετρήσιμη θα πρόσθετα εγώ. Και εδώ έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό και το γνωρίζετε. Επειδή είμαι φιλελεύθερη, πιθανώς δεν θα συμφωνήσω ποτέ με κάποιον από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και αυτό είναι ίσως το μόνο που μας χωρίζει. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση της καλής ποιοτικής ε, προσφοράς. Γιατί εγώ ως φιλελεύθερη αυτό το θεωρώ πάρα πολύ υποκειμενικό. Ποια είναι η καλή ποιοτική προσφορά στην εργασία, στην, στην ε, άσκηση, στη μαθητεία. Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, από τις καταστάσεις, τα προσόντα, τις δεξιότητες, ακόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έχω πρόβλημα με αυτή την καλή ποιοτική προσφορά, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μετρήσιμη. Και από τη σκοπιά της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα να το μετρήσουμε αυτό. Και είναι πραγματικά κάτι πολύ υποκειμενικό και ατομικό. Ίσως θα μπορούσε να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς το μετράς αυτό, την ποιότητα. Και ε, τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να ε, προχωρήσουμε προς αυτούς τους μετρήσιμους στόχους. Και ένα τελευταίο σας ευχαριστώ πολύ που αναφερθήκατε στην αναντιστοιχεία δεξιοτήτων και ε, θέσεων εργασία. Το συζητούμε και στην Επιτροπή Γυναικών αυτό εντατικά και μάλλον και στην ε, διάσκεψη που θα γίνει στις 10 Μαΐου. Αυτή η αντιστοιχία πραγματικά είναι τεράστιο πρόβλημα για την απασχόληση των νέων και θα πρέπει να αρχίσει να μας απασχολεί και μας πάρα πολύ νωρίς. Γιατί κάνουμε αλλαγές στην παιδεία, ε, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται αύριο, φαίνονται μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή αυτά που συζητάμε τώρα μην περιμένουμε έχουν αύριο αποτελέσματα, θα περάσουν χρόνια για να υλοποιηθούν. Σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομερείς ε, στατιστικές, αριθμητικά στοιχεία και όλες τις γραφικές παραστάσεις. Σας ενθαρρύνω να ασχοληθείτε περισσότερο με αυτά τα θέματα, όπως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες στην εφαρμογή όλων αυτών των προγραμμάτων για την απασχόληση των νέων γιατί χωρίς τεχνική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τοπική αυτοδίκηση δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρει. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή μας, τον Τέρεκ. Frau Kollegin bitte. συνάδελφος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ τον Σαν για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει αυτό το πολύ λεπτό θέμα και για μας και για το Κοινοβούλιο εν γέννη. Πράγματι με το Ταμείο Εγγύης για την Νεολαία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων, όχι μόνο στις χώρες του Νότου, αλλά γενικότερα. Αν δείτε τι ποσοστά ανεργίας έχουμε για τους ε, νέους ε, που και κάτω, ε, βλέπετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ε, άλλων ηλικιών εργαζομένους ε, ή κοντά τέλος πάντων, πολύ κοντά στο όριο, κοντά στην αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά ανεργίας των κάτω των 30. Και υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα, η σχολική αποτυχία κτλ. κτλ. Θα ήθελα να στηρίξω πολλέ προτάσει και τώρα με τον κύριο Βον, ιδίω σε ό,τι αφορά το πολύ εύστοχο και το είδαμε και με την εκπρόσωπο πριν του ελεγκτικού συνεδρίου των προτάσεων. Πολλές φορές οι εκθέσεις ε, ε, κατατίθεται γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα. Και μετά αλλάζει συγκυρία. Και δεν βλέπουμε με την έκθεση να αντικατοπτρίζεται ακριβώς το τι έχει γίνει με τα προγράμματα, με την εξέλιξη των ταμείων και το πώς έχουν τα κονδύλια κτλ. Αυτό είναι σημαντικό. Το ελεγκτικό συνεδρίο λοιπόν νομίζω θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη. Ένα τόσο σοβαρό και τόσο ε, εκτεταμένο φαινόμενο όσο είναι η ανεργία των νέων και κάτω των 30 είναι φυσικά ανάγκη να αντικείμενο μια ειδική έκθεση. Έχουμε διάφορα προγράμματα. Μάρκο Πόλο κτλ. Τέλο πάντων, πάντα πρέπει να έχουμε πρόβλημα στο πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που προστίθεται όταν συζητούμε πάντα ε, στο πέστη Κομισιόν για τους νέους, θα πρέπει να εμβαθύνουμε στον προβληματισμό μας γιατί βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται προσπάθειες ε, να εφαρμοστούν ε, κάποιες επιτυχημένες φόρμουλες ε, σε συμμεμονωμένα κράτη-μέλη και να εφαρμοστεί γενικευμένα αυτό. Όπως με την εγγύηση για την νεολαία, να εφαρμοστεί το διπλό εκπαιδευτικό σύστημα, το γερμανικό, σε όλες τις χώρες. Όμως αυτό ε, κάπως θέλουμε τέλο πάντων να πετύχουμε το εξή. Οι εργαζόμενοι, οι εργοδότε, οι επιχειρηματίε να δεσμευτούν ότι θα προσλάβουν ε, κάποιου οι οποίοι έχουν βγει από μια περίοδο μαθητεία ή από τι πτώσει κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά να αντιγραφεί το γερμανικό σύστημα. Να πάρουν α, ε, την ευθύνη για του εργαζόμενου εργοδότε. Αυτό δεν συμβαίνει όμω στην Ισπανία, τι άλλε χώρε του Νότου και σε πολλέ άλλε χώρε και με τις σχολές δεύτερης ευκαιρίας το ίδιο συνέβη ένα πολύ καλό ισπανικό ε, μοντέλο για νέους που είχαν αποτύχει στο σχολείο τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία αλλά τελικά σκοτώσαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα που είχε δουλέψει πολύ καλά στην Ισπανία προσπάθησε να το ε, αντιγράψουμε σε άλλες χώρες να το αναπαραγάγουμε και αυτό πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να προσπαθούμε να γενικεύσουμε προγράμματα που μπορεί για μια χώρα να είναι πάρα πολύ κατάλληλα αλλά πρέπει να έχουν υπόψη όλο το, το πρόγραμμα και τις λεπτομερίες του για να μην καταλήξουμε σε παταγώδει αποτυχίες σε άλλα κρατημέλη. Σε ό,τι αφορά για αυτούς τους νέους που δεν έχουν απασχόληση, ή θέση, πρέπει να δούμε τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε την εγγύηση για την νεολαία, έχουμε τον ορίζοντα 2020, έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προσφέρουν όλοι αυτοί, ε, όλα αυτά τα προγράμματα, θέσει εργασία ή ε, μαθητή. Θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βον για τα σχόλιά του. Πάρα πολύ επιτυχημένα, πολύ εύστοχα. Και νομίζω ότι και το ελεκτικό συνέδριο αλλά και η Κομισιόν θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Ευχαριστώ, συνάδελφος Τσέλερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς το συντονιστή του ΕΛΚΟ και σκιώδη κύριο Σάρβαμα να το δικαιολογήσω που δεν μπορεί να είναι εδώ. Μου ζήτησε να σας μεταφέρω τις δικές του παρατηρήσεις ο συνάδελφος από το ΕΛΚ σε σχέση με αυτό το έγγραφο εργασίας αλλά στα αγγλικά το κείμενό του. Δεν το μετέφρασα στα γερμανικά. Θα προσπαθήσω με τα αγγλικά που έχω μάθει από το σχολείο να σας το διαβάσω. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για την ε, έκθεση του που είδε πάρα πολύ ενδελεχώ το θέμα και έχει καταθέσει και σημαντικέ συστάσει για μελλοντικά μέτρα. Επίση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή κύριο Βόν για την καλή δουλειά που έκανε με το έγγραφο εργασία του και με το οποίο συμφωνούμε, όπω και με τι προτάσει του. Η εγγύηση για την νεολαία και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχουν στόχο τη μείωση τη ανεργία των νέων. Αλλά είναι κάπω απογοητευτικά τα αποτελέσματα τι θα περίμενε κανείς από ένα πρόγραμμα με περιορισμένους πόρους. Περίμενε ε, αντίστοιχα να έχουμε μεγάλα προβλήματα. Με τις ε, έκθεση του λεκτικού βλέπουμε ότι δεν έγινε δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τελικά της ανέργειας των νέων ε, σε όλη την Ευρώπη. Αρεσιμότητα, οι χρονικοί περιορισμοί, δεν δόθηκε ε, και τη έμφαση στι τέσσερι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ε, και να τα λέμε υπόψη ε, στη χάραξη μελλοντικών μέτρων. βέβαια, υπήρξαν και πολλέ επιτυχίε για τι οποίε είναι υπεύθυνη η εγγύηση για του νέου και πολλοί νέοι θα επωφεληθούν για τα πολλά επόμενα χρόνια από αυτό το πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι νέοι και Ευρωπαίοι, οποίοι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν να, να ενηλικιώνονται ε, χωρίς να έχουν καμία εμπειρία επαγγελματική και χωρίς να έχουν ε, επαρκή ε, προσόντα για να μπορέσουν να βρουν μια θέση εργασίας. Ε, θα... Είναι λοιπόν περιορισμένες οι δυνατότητές τους να, να κατακτήσουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Αν πραγματικά το εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει να δώσει προτεραιότητα στην ε, απασχόληση των νέων, θα πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες ε, για να βρει ε, κατάρτιση και θέση εργασία για του νέου. Και η Κομισιόν και τα κρατημένα θα πρέπει να αυξήσουν τι προσπάθειε και να συνεχίσουν να στηρίζουν την εγγύηση για την ολέα. ενέργεια. ανεργία των νέων θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και από πολιτικής πλευράς και από οικονομικής πλευράς. Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ποιοτικές θέσεις εργασίας, στην επιχειρηματικότητα είναι προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν η απασχόληση των νέων να γίνει σημαντικός πυλώνας ε, του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Αυτά λέει ο Πίτερ Σάρβαμα και ευχαριστεί όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νόβακοφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ την κυρία την κυρία Ιβάνοβα για, ένα, για μια εξαιρετική έκθεση επί ενός θέματος που είναι πολύ σημαντικό και που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα συμφωνούσα τους με την Μαρτίνα για την πολύ καλή ποιότητα και θα έλεγα ότι πέρα των διαφορετικών περιφερειών και χωρών Ακόμα και για διαφορετικούς ανθρώπους η ποιότητα σημαίνει κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν στο μέτρο του δυνατού να βρίσκουμε μια ατομική προσέγγιση ώστε ένας άνθρωπος να βρίσκει μια βιώσιμη απασχόληση. Αλλά μόλις πριν από μία εβδομάδα ψηφίσαμε να αυξήσουμε τον προεπολογισμό της πρωτοβουλίας για τους νέους. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετα κονδύλια. Και επομένως μιλούμε για πολύ συγκεκριμένη κατανομή του προϋπολογισμού και πολύ σημαντικό κονδύλι, αλλά πρέπει να συνεισφέρει με ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η επιδότηση μπορεί και να είναι μία οδός για κάποιες περιπτώσεις, ίσως, αλλά πέραν αυτού θα πρέπει να προσεγγίσουμε τους εργοδότες ώστε να παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εργαζομένους. Πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι έχουμε υψηλότατη άνευ προηγουμένου ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν εργοδότες που δυσκολεύονται ιδιαίτερα να βρουν ανθρώπους, υπαλλήλου με κατάλληλες δεξιότητες, με κατάλληλα προσόντα. Πρέπει λοιπόν να κατευθυνθούμε προς τους νέους ανθρώπους εκείνους που θέλουν, που έχουν τις δεξιότητες και θέλουν να διεχετευθούν στην αγορά. Στη Γερμανία έχουμε την, την, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας και τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης ειδικών και αναλυτών στην αγορά. Και ίσως αυτό το μοντέλο πρέπει να το υιοθετήσουμε περισσότερο γιατί δίνει αποτελέσματα. Θα πρέπει βέβαια να παραδεχθεί κανείς ότι σε κάποιες χώρες οι παραδόσεις είναι διαφορετικές και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παντού την ίδια προσέγγιση. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να παράσχουμε στήριξη στους εργοδότες να προσλαμβάνουν και κυρίως να εκπαιδεύουν συνεχώς τους εργαζομένους τους. πολύ συχνά μου λένε ότι είμαι μόνιμος εισηγητής για θέματα ανεργίας στην νεολαία. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι μόνιμος ενδιαφερόμενος, δηλαδή ασχολούμαι μονίμως με το θέμα αυτό. Είναι κρίσιμη σημασία πιστεύω και νομίζω ότι και η κυρία Ιβάνοβα ασχολείται εξίσου ενεργαμεμένα και η έκθεσή της είναι εξαιρετική. Oui, madame euh, la présidente. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου. Κύριε Ζακ, θέλω να συγχαρώ την κυρία Ιβάνοβα και το ελεγκτικό συνέδριο για την ποιότητα τη έκθεση. Όπω είπαν και προλαρίστατε συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μα τον κύριο Βόν. Εμένα κάτι μου λείπει μόνο, έχω ένα παράπονο. Σε ένα συγκεκριμένο και τόσο σημαντικό θέμα για τους ε, Ευρωπαίους νέους, να είναι τόσο άδεια τα έδρανα εδώ. Εγώ είμαι ευγενή, δεν θέλω να κατηγορήσω τους απόντες, αλλά θα επιθυμούσα ο συνάδελφος Φλάναγκαν να έχει επιδείξει τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο ενθουσιασμό ε, και το ίδιο στένος που ε, ανέπτυξε προηγουμένως σε σχέση με την εσωτερική πολιτική της Ουγγαρίας. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι οι Ιρλανδοί ε, άνεργοι νέοι ε, παθιάζονται για την εσωτερική εγκροκή πολιτική. Ε, ωστόσο, ένα πράγμα γνωρίζω, του ενδιαφέρει πάρα πολύ το στένος με το οποίο υπερασπίζονται τα δικά τους μελήματα οι προβουλευτές τους ειδικά σε μια χώρα που αγγίζει το 20% η ανεργία των νέων. Ευχαριστώ. Εδώ τελειώσαν ε, οι τοποθετήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο έχει ο κύριος Ούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ευχαριστήσει το λεκτικό συνέδριο για την έκθεση αυτή. Βεβαίως σημειώσαμε με μεγάλη προσοχή τα όσα ε, περιγράφει. Μπορούμε να δεχτούμε κάποιες συστάσεις, αλλά δεν συμφωνούμε με το βασικό συμπέρασμα ότι η ε, ε, πρωτοβουλία για την νεολαία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και ήταν περιορισμένη η συνεισφορά της. Θέλω να κάνω κάποια γενικά σχόλια. Αν θέλετε πριν ανάλυση, διαβάστε μας. Η εγγύηση για την νεολαία είναι πραγματικότητα πλέον στην Ευρώπη με εκατομμύρια ε, νέους να εγγράφονται για να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα και να λαμβάνουν προσφορές. Ακούσαμε ότι η ανεργία των νέων μειώθηκε ε, κατά 1,7 εκατομμύρια. Είναι μια ε, ολοκληρωμένη και μεγάλη μεταρρύθμιση αυτή και χρειάζεται ε, καιρό για να αποφέρει καπού και πολλά από τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται η εκθεσή σας ε, ανάγονται στο 2014-2015 στην αρχική εφαρμογή του σταδίου αυτού μάλλον στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής του συγκεκριμένου ε, μέσου στα κράτη-μέλη έχει προχωρήσει από το 2016 και μετά η εφαρμογή και η πρωτοβουλία για την νεολαία ανταποκρίνεται στο ρόλο της και κυριαρχεί στις πολιτικές αποφάσεις ε, η υλοποίηση αυτής στις επιλέξιμες χώρες. Οπότε τα αποτελέσματα για την πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να ε, θεωρούνται προκατακτικά, γιατί πάντα μεσολαβεί κάποιος χρόνος και υπάρχει διαφορά φάσεως από τη στιγμή ε, της έκθεσης μέχρι τη σημερινή κατάσταση. Γιατί η έκθεση αναφέρεται σε στοιχεία του παρελθόντος. Τώρα, ε, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση. Είναι σωστή η χρηματοδότηση, λείπουν πόροι, ρωτάει το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρωτοβουλία ε, για την νεολαία δεν είναι ε, η μόνη πηγή χρηματοδότησης 6,4 δις ήταν η αρχική ε, αυξήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 1,2 δις την περασμένη εβδομάδα. Είναι πολύ ισχυρό μέσο χρηματοδότησης λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την εγγύηση για την νεολαία. Γνωρίζουμε ε, από την Eurofund και το ILO που έχουν κάνει Μελέτε ότι χρειάζεται να συμπληρώνονται όλα αυτά από εθνικού πόρου. δεν αρκούν μόνο οι ευρωπαϊκοί. Ένα άλλο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι η εγγύηση για την νεολαία δεν έχει να κάνει μόνο με αριθμού, αλλά με διαρθρωτικέ αλλαγέ και πολύ περισσότερα για ε, βελτίωση της μετάβασης από το σχολείο στην αγορά εργασίας, για τα εκπαιδευτικά συστήματα, πρέπει να στηθούν συστήματα μαθητείας, θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζουν τους νέους οι κρατικές δομές απασχόλησης, υπηρεσίες δηλαδή κρατικές. Απαντώ σε δύο ερωτήσεις του εισηγητή για τις βελτιώσεις που έχουν γίνει από την ε, ημερομηνία της έκθεσης. Σας είπα για την πρωτοβουλία αυτή, τα στοιχεία βελτιώνονται αργότερα τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τα χρόνια στα οποία αναφέρεται η έκθεση. Συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη, ε, οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Στην Κροατία έχουμε ένα νέο σύστημα καταγραφής, στη Φιλανδία μια μόνο απευθυντική θηρίδα ή ένα νέο τρόπο υπολογισμού και εντοπισμού στη Γαλλία ε, για τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την αποφύτισή τους. Τώρα παρακολουθούμε και την ποιότητα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Έχουμε και άλλο τρόπο παρακολούθησης με κάποιους δείκτες παρακολούθησης follow-up ε, εντός ενός πλαισίου δικτών. Να δούμε. Ένας νέος που δέχτηκε μια τέτοια προσφορά, πού βρίσκεται μετά από 6, 12 και 18 μήνες για να καταλάβουμε αν ήταν ποιοτική η προσφορά. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι η καλή ποιοτική προσφορά σημαίνει μόνιμη και βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας. Ακούμε όμως την έκκληση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το ε, Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που μας ζητούν να εξακολουθούμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή την ποιοτική και θα δούμε τα ποιοτικά πρότυπα για ε, τις προσφορές αυτές αρχές Μαΐου. Πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να απαντήσω και στα όσα είπε το ελεγκτικό συνέδριο για την ευθύνη υλοποίηση αυτή τη πρωτοβουλία ε, για τι εγγύηση για την νεολαία. Είναι σαφέστατη αυτή η ευθύνη των κρατών μελών. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή και την υλοποίηση αυτών των σχημάτων και των πρωτοβουλειών μέσω τεχνικής αρρωγής, ε, δημιουργίας δυνατοτήτων και διδασκόμενοι ένας από τον άλλον, όπως ακούσαμε προηγουμένως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ιβάνοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις ε, παρατηρήσεις τους ε, και τα σχόλιά τους. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια τους. Θα ξεκινήσω υπογραμμίζοντας ότι αυτό που ήταν και είναι για μας καινοτομία του εγγυητικού μέσου για τους νέους και για να επανέλθω στο θέμα των προσδοκιών γιατί εκεί δεν τα καταφέραμε. Εδώ ο στόχος ήταν συστηματικά να προσεγγίσουμε όλους τους νέους, όχι μόνο εκείνους που ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή μαθητείας, εντός τεσσάρων μηνών. Επί τη βάση των μεγεθών που αναλύσαμε στην έκθεση, αυτός ο στόχος δεν έχει καλυφθεί, δεν έχει επιτευχθεί. Και η Κομισιόν στη Λευκή της Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης λέει ότι υπάρχει αναντιστοιχεία μεταξύ των προσδοκιών και των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις καλύψει. Επομένως αυτό υπογραμμίζει απλώς το ίδιο το συμπέρασμα της Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε να λειτουργήσει καλά το εγγυητικό μέσο για τους νέους. Δεν φαντάζομαι ότι κανείς από τους ομιλητές δεν θα επιθυμούσε κάτι τέτοιο. Όλοι επιθυμούμε να τα καταφέρει. Και οι που παρατηρήσαμε κατά και του ελέγχου είναι αδυναμίες που τις υποβάλλουμε προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά. Να βελτιωθεί το σύστημα και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Τώρα μια πολύ σημαντική ερώτηση έγινε από τον κύριο Βάλλη και την κυρία Αγιάλα ε, σχετικά με τους σπόρους ήταν ένας κίνδυνος τον οποίο υπογραμμίσαμε από την πρώτη έκθεση σχετικά με το εγγυητικό μέσο ότι δηλαδή η χρηματοδότηση ήταν ελλειπής ε, σύμφωνα με εκτιμήσεις ανεξαρτήτων φορέων όχι του ελεκτικού συνεδρίου ο ILO που λέει ότι το ετήσιο κόστος για της εγγύης αυτής ήταν 45,4 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος. Η Eurofound βρήκε 54 δισεκατομμύρια. Και γνωρίζουμε ποια είναι η χρηματοδότηση συνολικά του εγγυητικού μέσου. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν έλλειμμα, mismatch για να συνενούμεθα. παρουσιάστηκαν μια σειρά από μέτρα για να χρηματοδοτηθούν, αλλά κανένα κρατος δεν μπορούσε να υποβάλει ένα, μια εκτίμηση κόστους του, για, του συνόλου των αναγκών για τέσσερις μήνες. Προφανώς και δεν μπορεί λοιπόν το μέσο αυτό να απευθυνθεί στο σύνολο του πληθυσμού. Εντός της υφιστάμενης χρηματοδότησης, χωρίς εμείς να λέμε ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη η χρηματοδότηση, υπάρχει αναντιστοιχεία μεταξύ των προθέσεων και της χρηματοδότησης που διατίθεται. Επίσης έγινε μια ερώτηση από την κυρία Γιάλα σχετικά με τη χρονική στιγμή της έκθεσης και συμφωνώ απολύτως μαζί σας πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι. Οποιαδήποτε ειδική έκθεση πρέπει να την υποβάλουμε εντός του πιο σύντομου χρονικού διαστήματος που θα ήταν δυνατόν. Για την προηγούμενη εγγύηση είχαμε κάνει 10 μήνες, για αυτήν εδώ λίγο παραπάνω. Ελέγχθη επίσης ότι τα δεδομένα ίσως να είναι λίγο παλιά όχι απολύτως επικαιροποιημένα. Εκεί που είχαμε προσπαθήσει να ακολουθήσουμε μια εξάντε προσέγγιση ήταν για το πρώτο εγγυητικό μέσο. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτά που είχαμε υπογραμμίσει ε, πραγματοποιήθηκαν. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαμε ήταν τα τελευταία δεδομένα ΕΜΚΟ που είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη χρονική στιγμή, αλλά με την ευκαιρία, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή την όλη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των γενικών διευθυντών, των τμήματων. Αντιλαμβανόμαστε διάφορους περιορισμούς νομικούς και άλλους ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις συστάσεις και τις προτάσεις μας αυτές, διότι η κοινή μας ευχή και επιθυμία είναι να βελτιώσουμε το εγκαιρικό μέσο. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν, ευχαριστώ και τα κράτη-μέλη και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Άρα υπάρχει έτσι πασχαλινή ειρήνη ο εισηγητής για να Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Νομίζω και ελπίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι ήταν χρήσιμες εγγύσεις για την ΟΛΕ. Για να περιοριστεί το σκάνδαλο της ανέανικης ανεργίας στην Ευρώπη. Ας συμφωνούμε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος της λύσης εγγύσης για την ΟΛΕ. Τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλη ευθύνη και πρέπει να υλοποιήσουν δομές για να αξιοποιήσουν τις για την νεολαία και τις σχετικές ενισχύσεις και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το σημαντικότερο δε έχουν ευθύνη τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση της ανηρίας των νέων. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική προτεραιότητα. Είναι κατεπήγον αυτό. Αυτή είναι η δική μα προτεραιότητα και θα κάνουμε ό,τι το δυνατό για να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και ο ιδιωτικό τομέα έχει ευθύνη. Και αυτό που λέτε για τι καλές ποιοτικέ προσφορές, γιατί ακούστηκε αρκετέ φορέ. Αυτό που δεν θέλουμε σίγουρα είναι οι προσφορές είναι να τους βάλουν τους νέους να κάνουν φωτοτυπίες και να φτιάχνουν καφέ και τσάι. πρέπει να υπάρχουν και πια κριτήρια προσφορές που υποβάλλονται σε αυτούς τους νέους για, για μια θέση εργασίας. Δηλαδή να υπάρχει μια επαρκής και αξιοπρεπής αμοιβή και να τους παρέχει αυτή η θέση ε, κάποια ευκαιρία, κάποιες ευκαιρίες να βρουν μια καλύτερη θέση εργασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εν κατακλείδη όλοι συμφωνούν ότι αργά ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε αργά, ε, μπορούμε να το συζητήσουμε, υπήρχαν καθυστερήσεις, αλλά τώρα νομίζω ότι υπάρχει πρόοδος, εγγύες για την ολέα, συνολικά θέλουμε να συνεχιστεί έτσι να υπάρξει πρόοδος και σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις στο ελεγκτικό συνεδρίο είναι όλες χρήσιμες γιατί επισημαίνουν ζητήματα, επισημαίνουν προβλήματα του παρελθόντος από τα οποία μπορούμε όλοι να διδαχθούμε. Και ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον το πρόγραμμα για τον εγγύσεων γιατί η νεολαία. Έχει πολλά να προσφέρει για να απειλήσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας πω για τα επόμενα σημεία ότι δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το 10 και 11. Ε, άλλως έπρεπε να είχαμε οργανωθεί. Άρα θα ολοκληρώσουμε την ημερήσια διάταξη με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. και συγκεκριμένα τι νέε ρυθμίσει χρηματοδότηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμια Τράπεζα και τι επιπτώσει του προπολογισμό. Το συζητούμε γιατί είχαμε κάποιε εξελίξει. Ο πρόεδρο επεξελέγει στην ε, Παγκόσμια Τράπεζα, το διαπραγματεύτηκε. Έχουμε αποφασίσει δύο επιτροπών από τι 12 Απριλίου 2016. Έχουμε δύο αποφάσεις Κομισιόν, 2210 και 2250. και θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία ε, περί πρόκειται. Με την αναθεώρηση ε, των χρηματοδοτικών αρχών, funding principle, ε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σχετικά με την Παγκόσμια Τράπεζα. Από το 2014 υπάρχει μια χρηματοοικονομική συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το 2016 με τις αποφάσεις της Δίας Κομισιόν άλλαξε αυτή η συμφωνία. Πού είναι αυτές οι αλλαγές, τα καταπιστεύματα που ε, διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα, θα περιοριστούν τα, τα τέλη, τα διοικητικά, θα ήθελα να σας πω ότι για τα πρώτα 15 εκατομμύρια για τα ε, πρώτα 50 μειώνονται και για τα επόμενα 45 ε, μειώνεται ακόμη περισσότερο. 3% και 2% αντίστοιχα. Αλλάζει δηλαδή η κατάταξη. Καταποκοπή είναι λοιπόν αυτό 5,5% αφορά όλα τα καταπιστεύματα ε, που είναι αποδέκτες και διοργανώνουν ε, και μετά η μεγάλη μάζα δηλαδή και μετά μια άλλη εξειδίκευση τα καταπιστεύματα που ε, διεκπεραιώνει η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα και εδώ υπήρχε μια ενδιαφέρουσα συμπλήρωση, το 17% το κόστος ε, για το προσωπικό το παίρνει η Παγκόσμια Τράπεζα κάτω από Αυτό το 17% μου φαίνεται πολύ ψηλό και αφορά ε, ορομίσθιο, το προσωπικό που πληρώνεται με την ώρα και οι σύμβουλοι. Και αφορά αυτό όλα τα επίπεδα του management, γιατί δεν αναφέρει ποτέ ότι πρόκειται για εκείνους που εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο έργο και πληρώνονται με την ώρα. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακαλώ να την απαντήσει. Το έγγραφο λέει ότι έτσι αυξάνεται ε, το ποσοστό της τράπεζας από 5,47% σε 5,58% για την διεκπαιρέωση, αλλά θέλουμε ανάλυση αυτή με ευρώ και σέντς. Ε, εγώ προσπάθησα πάρα πολύ και κόπιασα για να καταλάβω τι λένε τα διάφορα έγγραφα και περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις από όλα αυτά τα πράγματα για ε, καταπιστεύματα που δρούν ε, σε επίγουσες ε, καταστάσεις και τι γίνεται μετά την απολύτως επίγουσα κατάσταση. Τι συνέχεια δίνεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει, γι' αυτό κάνω τέτοια εκτενή εισαγωγή, είναι τι αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αλλαγή αυτή. Στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερα καταπιστεύματα για οτιδήποτε ε, από ό,τι έχουμε σήμερα. Αυτή η εξέλιξη μας περιμένει και επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες από όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μου έχει εξηγήσει με διάφορες περίπλοκες ε, εξηγήσεις και υπολογισμούς ε, ότι θα μειωθεί σημαντικά το κόστος. Άρα τι σημαίνει ότι πληρώναμε υπερβολικά, μπορείτε να μας δώσετε ε, ένα κατάλογο για όλα τα multi-donor trust funds που έχουμε καταβάλει υπερβολικά ποσά. Αυτά συνοπτικά. Το βρήκα πάρα πολύ περίπλοκο, όσο και αδιαφανέ και πολύ θολό και συγκεκριμένο όλο αυτό. Και ρώτησα γιατί ισχύει κάτι τέτοιο και αυτό με απασχολεί. Αν δούμε όλες αυτές τις αλλαγές, καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον θα διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο η Παγκόσμια Τράπεζα από ό,τι μέχρι σήμερα. Και τι γίνεται με τους άλλους αποδέκτες, άλλους δικαιούχους, άλλων διεθνών οργανισμών ε, ορίσατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε μέσα στο λόγο, κύριε Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μια συμφωνία με την Παγκόσμια Τράπεζα το 2001, ε, χρονή συνεργασία, το 2014 έγινε μια μείζων αναθεώρηση του πλαισίου, το είπατε και εσείς, και έπειτα χρειάστηκε να δεχθούμε μια διάταξη που περιλάμβανε ρήτρα αναθεώρησης η οποία εφαρμόζεται και ισχύει για όλους τους δεπτές της Παγκόσμιας Τράπεζας και σχετίζεται με τη θέσπιση από την Παγκόσμια Τράπεζα μιας νέας πολιτικής ανάκτησης ε, καταστευμάτων που αναφέρατε κι εσείς. Αυτό, ε, αυτή η νέα πολιτική ανάκτηση υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, 30% του ε, μεριδίου το έχουν είπα, μετά ε, εφαρμόστηκε προοδευτικά στις συμφωνίες που έχει με άλλους οργανισμούς η Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η νέα πολιτική ανάκτησης κόστους είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε ε, έξωθεν, είναι μια στέκη απόφαση. Αλλά το σύστημα είναι πολύπλοκο, ήταν αρκετά απλό, 5% κατά αποκοπήν της Συμβουλής της Ένωσης τώρα περνάει σε ένα άλλο πολύπλοκο σύστημα με δύο διαφορετικά τέλη, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, προοδευτικά μειούμενα από 5 φτάνουμε στο 2% αλλά αυτή η φθήνουσα, αναδρομικο... προοδευτικότητα έχει να κάνει με όλο το ποσό, όχι μόνο με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι δίνεται ένα σημαντικό κίνητρο στην Ένωση και σε άλλους οργανισμούς να προσχωρήσουν σε μεγάλα καταπιστεύματα που να δημιουργηθεί έτσι η οικονομία κλίμακας. Έχουμε αυτό το τέλος επίσης 17% για το προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μόνο για το προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Άρα δεν εφαρμόζεται σε συμβασιούχους, επιχειρήσεις. Μιλάμε για τους παλίους της τράπεζας μόνο. 17% λοιπόν αυτό το τέλος. Και εφαρμόζεται μόνο σε ένα περιορισμένο τμήμα ε, των εισφορών προς την Παγκόσμια Τράπεζα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Όπως λέμε και στο έγγραφο που σας δώσαμε, έχουμε τα δύο άκρα, δύο παραδείγματα. Κάποια καταπιστεύματα για αγροτικά προϊόντα, όπου έχουμε μόνο το 2% της ε, εισφοράς για το προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και το 17% λοιπόν αυτό εφαρμόζεται στο 2% της εισφοράς. Άρα υπάρχει ένα γενικό τέλος λιγότερο από 5%. 4,59. Ένα άλλο ακραίο παράδειγμα. Δεν εφαρμόζεται κανένα τμήμα του καταπιστέματο από τρίτες χώρε μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα, προσωπικό τη παγκόσμια Τράπεζας, άρα μεγαλύτερη η επίπτωση, ο αντίκτυπος και εδώ έχουμε το Extractive Global Program Support. Έχουμε 2% ποσοστό του κόστους τη συμμετοχή τη συνολική για το προσωπικό και εδώ εφαρμόζουμε το 17% ακριβώς σε αυτό το, μάλλον όχι 22%, σε αυτό το 22%. 3,83 δηλαδή τελικά είναι το ποσό, γύρω στο 4%. Το 17 το εφαρμόζουμε στο 22 όπως είπα 100. Βλέπετε λοιπόν ε, τη διάκριση. Έχουμε ε, τα δύο αυτά παραδείγματα και στις δύο περιπτώσεις, είτε την, και στην έχει η, τη διαχείριση παντός τράπεζα, είτε κάποιο τρίτο μέρος, πάντα είμαστε σε καλύτερη πλέον θέση, σε καλύτερη κατάσταση με αυτή τη νέα ρύθμιση. Έχουμε ζητήσει στο πλαίσιο στρατηγική για την Ευρώπη 2020 ε, αναλύσεις και μελέτες από την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχουμε δει ποια είναι τα προβληματικά ε, καταπιστεύματα. Ξέραμε ότι με αυτή την αύξηση 17% για το προσωπικό θα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε συμφωνήσει με αυτή την ε, συμφωνία. Έχει τεθεί σε ισχύ αυτή η νέα πολιτική ανάπτυξη κόστο εδώ και μισό χρόνο και παρακολουθούμε πολύ κοντά τα πράγματα και βλέπουμε και μπορώ να σα επιβεβαιώσω ότι είμαστε κάτω από το 5%. Δηλαδή, είναι πιο μεγάλες οι οικονομίες σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Εμείς θα εφαρμόσουμε τη ρήτρα κεκτημένων δικαιωμάτων πάντως. Παναλαμβάνω, είμαστε κάτω από το 5%. Θα σας ενημερώσουμε για τα συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα με τα χρήματα που επενδύονται σε αυτά τα καταπιστεύματα. Είναι ένα απόλυτα διαφανές σύστημα, το επιβεβαιώνω αυτό. Θα πάρετε όλες τις ε, συμφωνίες για να δείτε ότι έχουμε τηρήσει τους κανόνες σε όλες τις περιπτώσεις με τα delegation agreements και θα γίνει και μία αποστολή 22-26 Μαΐου στην Παγκόσμια Τράπεζα που θα είναι και μια καλή ευκαιρία να δείτε και να ακούσετε από την Παγκόσμια Τράπεζα πώς εφαρμόζει αυτή τη νέα πολιτική. Και θα δείτε και τι άλλε ενέργειε έχουμε με την Παγκόσμια Τράπεζα σε σχέση με τα αποτελέσματα. Βλέπουμε επίση και τη δομή των λογιστικών ελέγχων και την πολύ αποτελεσματική διαχείριση συνολικά των καταπιστευμάτων. Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πιο πολύπλοκο σύστημα που μας επιβλήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και όχι μόνο σε εμάς, παραλαμβάνω σε όλους τους δωρητές. Εξίσου. Με τις διαπραγματεύσεις μας όμως νομίζω ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε ένα σύστημα που οικονομικά είναι πιο προσωφόρο για μας και μας δίνει δυνατότητα να σας ενημερώνουμε και καλύτερα για τα αποτελέσματα των πολιτικών. Αυτά είχα να πω και μπορώ βέβαια να απαντήσω και σε περαιτέρω ερωτήσεις. Yeah, Ευχαριστώ πολύ. Έχω ερωτήσεις για να απαντήσετε. Για ποιο λόγο λέτε ότι υπήρχε η δυνατότητα ε, να έχετε έκτακτες ρυθμίσεις για έκτακτες ανάγκες και τώρα το έχετε διαγράψει αυτό. Για ποιο λόγο. Δεν θα χρειαζόταν έτσι και αυτή η αλλαγή αφού η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να πάρει περισσότερα ακριβώς με τις ε, ρήτρες για την εξαίρεση. Μετά γίνεται μεγάλη ε, ε, έντονη συζήτηση στις συμφωνίες για τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα. Ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια χρήματα σε ένα ταμείο έτσι ώστε το καταπίστευμα να μπορεί να χρηματοδοτεί κάποια πράγματα που δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι επιλέξιμα. Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, δηλαδή που δεν το χρηματοδοτούμε εμείς και θα το χρηματοδοτεί το καταπίστευμα. Και μετά, πόσα trust funds της Παγκόσμιας Τράπεζας λειτουργούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί συνδέονται με στόχους του ορίζοντα 2020. Εγώ θα προτείνω σε τούτη την Επιτροπή και την Επιτροπή Προϋπολογισμών να μπλοκάρουμε το δρόμο προς τα trust funds, γιατί επικρατεί πλήρης αδιαφάνει ε, και πλήρες σκότος. Είναι ένας κομψός τρόπος και γρήγορος να δαπανούμε ε, χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νύψει τα σχήρα τη και τα ε, ρίχνει όλα στην Παγκόσμια Τράπεζα γιατί δεν τα διαχειρίζεται ίδια. Αυτός ο τρόπος αποκέντρωσης να φεύγουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έχω φανταστεί έτσι εγώ όταν τα ψήφιζα ως νομοθέτης για θέματα προπολογισμού έχουν ανάψει καμπανάκια εδώ για μελλοντική ε, εξωτερήκευση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει στην ΤΕΦΚΟ γιατί να έχω 5.000 υπαλλήλου όταν όλα τα αναθέτεται εξωτερικά και φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν είστε καν, δεν συμμετέχετε στη διαχείριση. Και μάλιστα βγάζετε την ώρα της απ' έξω κανονικά. Αυτά θέλω παρακαλώ μου πατήστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι στα έγγραφα που σας μεταδώσαμε υπάρχουν πλήρες πληροφορίες για τα καταπιστεύματα. Νομίζω 7 είναι αυτά επί των οποίων υπάρχει σημαντικότερος αντίκτυπος από την ανάκτηση. Έχετε πάντα στον πλήρη κατάλογο για το σχόλιο σας θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολος τρόπος για την Κομισιόν αυτός. Όταν κοιτούμε τα καταπιστεύματα τα οποία διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα, θεωρούμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να τα χρησιμοποιήσουμε. Να σας φέρω για παράδειγμα το Αφγανιστάν. Έχουμε σαφείς δείκτες τον αριθμό των, των παιδιών που έχουν πρόσβαση στα σχολεία ή των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, στην υγειονομική περίθαλψη κτλ. Δηλαδή δεν είναι χρήματα που δίνονται χωρίς να υπάρχει άλλη παρακολούθηση. Υπάρχουν τακτικές υποβολές εκθέσεων και προς εσάς και στην όλη διαδικασία dispatch παρακολουθείτε την αποτελεσματικότητα της όλης αυτής της διαδικασίας. Και γι' αυτό έχουμε όλη, όλο αυτό το πλαίσιο, ένα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης και επιτήρησης προκειμένου να και πρέπει να εξασφαλίσουμε φυσικά ότι ε, χρηματοδοτούμε τα, τα πράγματα που θέλουμε. Δηλαδή το κομμάτι του προγράμματος το οποίο έχουμε στοχεύσει. Ώστε στο τέλος διαδικασίας να είμαι σε, θέση να σας δείξουμε ότι αυτό το κομμάτι καλύπτεται από ε, επιλέξιμες δράσεις υπό την περίοδο τη δημοσιονομική χ και άπτεται, ε, έχει, σχετίζεται με μια χώρα με την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε ε, εταιρική σχέση αναπτυξιακής βοήθειας ή οτιδήποτε άλλο. Σε οποιαδήποτε στιγμή όμως αυτές οι συμφωνίες μπορούν να τερματιστούν. ώστε να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα δαπανώνται κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για στόχους που αποκλίνουν από τις αρχές μας, αν θέλετε. Για τις δε διατάξεις ε, εκτάκτου ανάγκης, που είναι σχετικά καινούργιες, σε κάθε περίπτωση έχουμε, ε, ε, επιτρέπεται η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συστήματα πολλαπλών δωρητών ώστε να έχουμε σημαντικό αντίκτυπο, να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι θετικός ο αντίκτυπος της βοήθειάς μας, όπως το κάναμε με το Αφγανιστάν. και για την σύσταση νέων καταπιστευμάτων πρέπει να μπορούμε να συνεισφέρουμε και Εκτός από αυτά που διαχειριζόμαστε εμείς, σε καταπιστεύματα που διαχειρίζονται άλλοι φορείς. Και θεωρούμε ότι πράγματι ο αποτελεσματικότερος και πιο αξιόπιστος ε, εταίρος στη ε, διαχείριση των καταπιστευμάτων αυτών είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο ερωτήσεις που έκανα και προηγουμένως, αλλά δεν απαντήθηκαν ακόμα. Το 17% για τα καταπιστεύματα που ε, ε, υλοποιεί η τράπεζα. Ποιο προσωπικό είναι αυτό, τι συμπεριλαμβάνεται εκεί. Είναι προσωπικό που εργάζεται στο συγκεκριμένο έργο ή φτάνει και μέχρι την κυρία Λαγκάρτ. Was ist die Auswirkung ε, ε, οι άλλοι οι δωρητές. Και γιατί είναι τόσο απόρριτο τώρα αυτά και γιατί τέτοια είχε μύθια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στα κείμενα. Α, και κάτι ακόμα. Το διαπραγματεύτηκε η αντιπρόεδρος. Η τότε αντιπρόεδρος τι συμμετοχή είχε σε αυτές τις συμφωνίες. No translation. Um, Ζητώ συγγνώμη, έχασα ένα τμήμα της ερώτησής της. Το 17% καλύπτει το προσωπικό που εργάζεται επί του προϊόντος. Στο παράρτημα, ή μάλλον συμφωνία πλαίσιο, έχουμε σχέδιο ενδεικτικού προϋπολογισμού που δείχνει ποιος εργάζεται σε τι προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι δεν χρηματοδοτούμε τίποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση που θέλετε. Για την Αντιπρόεδρο Γεωργίευα μπορώ να σας ε, βεβαιώσω ότι είχαμε τη συμφωνία αρχικά του 2014 και είχαμε και μια ρήτρα αναθεώρησης για όλους τους δωρητές. Ως συνέπεια της νέας πολιτικής ανάκτησης κόστους της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2015. Και σε καμία χρονική στιγμή ουδέποτε δεν λάβαμε οποιαδήποτε ένδειξη από το γραφείο της Αντιπροέδρου Όλα αυτά τα διαπραγματεύτηκε ο Γενικός Διευθυντής Προϋπολογισμού με τις αρμόδιες μονάδες της ΔΕΒΚΟ το οποίο το έχει ξαναπεί η Αντιπρόεδρος, το έχει επιβεβαιώσει. Η διέρεση αυτή εργασία ήταν αναπόφευκτη λόγω της πολιτικής ανάκτησης κόστους, επαναλαμβάνω, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Yeah. On Για άλλους δωρητές, αυτή είναι μια ερώτηση που θα σας ενθάρρυνε να την διαβιβάσετε στην Παγκόσμια Τράπεζα, διότι δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση, τη διαχείρισή τους άλλων δωρητών. Υποτίθεται ότι ισχύει η ίδια πολιτική για όλους και εμείς Πράγματι αυτό πιστεύουμε, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίε για τις ΗΠΑ ή άλλους σημαντικούς δωρητέ. Ε, αλλά εσεί μιλούσατε για σύγκριση με άλλους διεθνεί οργανισμούς. Ίσως και εκείνοι θα το βρίσκαν ενδιαφέρον, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, Πρόεδρε, Κοιτάξτε, εμείς έχουμε το ίδιο όριο, αυτό που προβλέπει ο, ο κανονισμός, 7% με όλους τους εταίρους και με τα Ηνωμένα Έθνη, με όλους τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η Παγκόσμια Τράπεζα λόγω της εκτέλεσης των δράσεων αυτών και λόγω των καταπιστευμάτων επιτυγχάνουν οικονομία κλίμακας μεγαλύτερη από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Διότι μια μόνιμη παρουσία επιτόπου όπως έχουν τα Ηνωμένα Έθνη θα απέρεε σε μεγαλύτερο κόστος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για διαφορετικές προσεγγίσεις με τις συμφωνίες αυτές καταρθώσαμε να περιορίσουμε συνολικά το κόστος των καταπιστευμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και οπωσδήποτε αυτό είναι πιο οικονομικό από το να είχαμε περιφερειακά γραφεία σε διάφορες χώρες στον κόσμο. Ευχαριστώ. Εμείς είμαστε μια επιτροπή που εξετάζουμε πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν. Ε, θα σα ήμουν ευγνώμων να μας δίνατε ένα κατάλογο με το τι έχουμε δαπανίσει, ποια είναι τα ποσά, ποιο είναι το ε, κόστος το διοικητικό του προσωπικού και όλα αυτά. Και να δούμε τι έχουμε ε, ε, καταβάλει και ποια είναι υπερβολικά. Και ρωτώ γιατί όσες αυτέ οι συμφωνίες είναι τόσο εμπιστευτικέ και απόρριτε. Οι αποφάσει Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι σήμερα δεν είναι δημόσιες προσβάσιμες. Για ποιο λόγο, ευχαριστώ. Ήδη απαντήσαμε στο ερώτημα αυτό ότι όλες οι αποφάσεις κομισιών που εγκρίθηκαν το 2016 είναι στο Μητρό με, από τότε που υπογράφηκαν. Είναι εκεί ακριβώς που μπαίνουν ε, όλα τα ε, έγγραφα της Κομισιόν. Δεν την κρύψαμε τη συμφωνία. Μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση τύπου ε, όταν υπεγράφει Άρα, από ό,τι ξέρω, δεν ε, τις κρύψαμε αυτές τις συμφωνίες. Και είναι στο δημόσιο μητρό των εγγράφων από τότε που εγκρίθηκαν αυτές οι νέες αποφάσεις. Ναι, this is not the case, believe me. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, πιστέψτε με. Προσπάθησα να τα βρω πραγματικά τα έγγραφα άφαντα. Πολύ σκληρά προσπάθησα. Να μας στείλετε το σύνδεσμο, το link τότε να το βρούμε. Ωραία, ολοκληρώθηκε το θέμα αυτό. Α, ο σύνδεσμος Σέλερ. Δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά αυτά που ακούμε εδώ και ακούμε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι η κατεξοχήν, ε, τράπεζα, ε, κατεξοχήν θεσμός που είναι πιο αποτελεσματικός στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Υπάρχουν και άλλοι που αμφιβάλλουν σφόδρα. Και αν δω πώς έχει η δομή και η διάρθρωση, εκεί δεν συμμετέχει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Κομισιόν, ούτε έχουμε δικαίωμα ψήφου σε αυτό το θεσμό. Και εκεί κάνουν κουμάντο κάποιοι άλλοι, πολύ διαφορετικοί. Και αν δίνουμε τόσα πολλά χρήματα που πρέπει να πάνε στην ε, αναπτυξιακή βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία και στηρίζουμε αυτό το θεσμό, θα πρέπει να έχουμε και περισσότερη διαφάνεια για το πού καταλήγουν αυτά τα χρήματα. Ακόμα και αν συγκεντρώνονται αυτά σε καταπιστεύματα, πολλές φορές αυτό είναι για συγκάλυψη διαφόρων μέτρων που εφαρμόζονται και να μην τα πολύ μαθαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, Πρόεδρος, και εγώ αυτό πιστεύω. Θα πρέπει να παραμείνουμε στο θέμα αυτό. Κύριε Βάλμπροκ, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Τσέλερ και να μας πείτε και τι σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς φαντάζεται τη μελλοντική συνεργασία της με την Παγκόσμια Τράπεζα για τα καταπιστεύματα και τα λοιπά ταμεία. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε άλλους εταίρους. Ε, εκφράζομαι προσεκτικά και επιφυλακτικά, ας με τον ΟΗΕ και άλλους εταίρους. Τώρα πρόκειται για την Παγκόσμια Τράπεζα. Ε, ε θα ήθελα να πω κάτι υπάρχουν κάποια έργα στα οποία διακρίνεται η Παγκόσμια Τράπεζα και είναι αποτελεσματική και ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους περιορισμούς. Έχουμε δημιουργήσει εμείς μια νέα πλατφόρμα η οποία δίνει πλήρη ενημέρωση ε, για τον αντίκτυπο των συνεισφορών, των δωρητών, τι τόπο πιάνουν τα χρήματα αυτά δηλαδή και Επίσης, ε, ε, ε, εργαζόμαστε συνεχώς προς την κατεύθυνση αυτή. Να είναι σωστή η πληροφόρηση και διαφανής και χρήσιμη και ωφέλιμη. Και έχουμε την, την προσέγγιση για το καλύτερο λόγο κόστους-οφέλους. Η Παγκόσμια Τράπεζα δεν είναι ο μοναδικός εταίρος μας για την αναπτυξή συνεργασία. Συνεργαζόμαστε και με τον ΟΗΕ και με οργανισμούς των κρατών μελών και όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για το κόστος και τη διαχείριση. Και είναι και πάρα πολύ λογικό. Δεν μπορούμε να αναθέτουμε σε κάποιον τρίτο ε, μια εργασία που βγαίνει πιο ακριβά από το να την κάναμε εμείς με αυτεπιστασία. And, and, and to complete the... και για να συμπληρώσω, θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε DEFCO με την DGNIR για να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου που δραστηριοποιείται και η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Και αυτό συνδέεται και με τη στρατηγική 2020, όπου έχουμε συνενώσει πολλές μελέτες σε ε, μια ενιαία προγραμματική μελέτη. Δεν βλέπω μείζονες αλλαγές ε, να έχουμε στο μέλλον με την Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά θα επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα και στη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό θα εξακολουθήσουμε να το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την προθυμία που που είχατε να έρθετε. Ολοκληρώνεται εδώ η δημόσια συνεδρίαση. Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα και στους διερμηνείς φυσικά και να περάσετε τις λίγες αυτές μέρες ξεκούραστα και μετά θα πάμε στην Πολωνία με μια μικρή αντιπροσωπεία. Είστε επανειδήν, καλά να περάσετε, χαίρετε.